Ladies and gentlemen, good morning, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Καλημέρα σα, αγαπητοί συνάδελφοι. Προσδεθείτε. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, wir haben Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα το πρωί έχουμε την ευχαρίστηση πολλές ψηφοφορίες να κάνουμε. Μπορεί να διαρκέσει πολύ αυτή η διαδικασία. Μπορεί όμως να πάει και πιο γρήγορα. Θα κάνω ό,τι μπορώ, ό,τι περνάει από το χέρι μας, να πάμε πιο γρήγορα. Αλλά μπορείτε και να με βοηθήσετε για να επιταχύνουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ξεκινάμε με πρώτη ψηφοφορία, το σημείο 13. Με την ασφαλή τροφοδοσία φυσικού αερίου. Έκθεση Βιντάλ Κουάντρα του συναδέλφου μας. Ξεκινάμε με την ψηφοφορία λοιπόν. Πρώτα έχουμε Πρώτα να δοκιμάσουμε ηλεκτρονικά. Εντάξει, μπορούμε να δοκιμάσουμε ηλεκτρονικά. Λειτουργούν όλα. Η πρώτη ψηφοφορία. Αν είμαστε ικανοποιημένοι είναι Αρχίζει, αρχίζει η ψηφοφορία να δούμε. Πέρας ψηφοφορίας. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι. Τι γίνεται με αυτό. Εδώ μπρο, έτσι. Εντάξει, οκ. Okay. εναντίον. Ποιο είναι αυτός. Ε, κάτι θα πρέπει να πούμε με αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πρώτη ψηφοφορία. Χωρί αστεία. Συμβιβασμός 13. Όσοι είναι υπέρ συμβιβαστικής πρότασης 13. Κατά. Αποχές. Ε, υιοθετείτε. Συμβιβασμός 14. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 1 υπέρ κατά αποχές υιοθετείται. Έτσι καταπίπτουν όλα στη συνέχεια. Μέχρι τον συμβιβασμό 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτουν όλα και δεν θα, στα, δεν θα σας τα διαβάσω καν. Και περνάμε στο συμβιβασμό 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε καταπίπτουν αρκετές σελίδες στη συνέχεια. Ωραίο αυτό με τους συμβιβασμούς. Συμβιβασμός 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 3α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε καταπίπτουν πάλι κάποιες σελίδες εκεί και περνάμε στην 141 τροπολογία. Τροπολογία 141 ως προσθήκη στο συμβιβασμό 3 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Περνάμε αμέσως στο συμβιβασμό 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Και πάλι κάποιες σελίδες γυρνάμε που καταπίπτουν. Συμβιβασμός 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Και ξεφυλίζουμε παρακάτω συμβιβασμός 6. Υπέρ. Συμβιβασμός 6. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Προχωράμε παρακάτω. Πολλές σελίδες είναι αυτές. Τι γίνεται εδώ. Συμβιβασμός 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Και συνεχίζουμε. Πολλές σελίδες. Σιγά σιγά για να τα προλάβουμε. Συμβιβασμός 9. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβασμός 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβαστική πρόταση 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Συμβιβαστική τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Και τώρα συνεχίζουμε εδώ, έτσι, επιμέρους ψηφοφορίες ξεχωριστές. 484 και 485 ταυτόσιμες υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν να ελέγξουμε. Πολύ ωραία. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Είναι ίσως καλύτερα. Ελέγχουμε. 484-485 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Ένα Ένας μη εγγεγραμμένος non-attached ε, ε, παραπάνω. Και τι γίνεται. Και ένας σοσιαλιστής. Και ένας από το ΕΛΚ. Μάλιστα. Ε, πολλοί είναι παραπάνω εδώ. Υπερβολικά πολλά μέλη παρόντα. Χωρίς μικρόφωνο η παρέμβαση. Εντάξει τώρα και η μη γραμμένη. Ένας παραπάνω πάλι. There are two members. Mr. Secretary, what's going on with this? Well, okay. It's okay. Εντάξει τώρα, πολύ καλά. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. 484-485 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 28 υπέρ 24 εναντίον εγκρίθηκε. 486 τροπολογία τώρα. Παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο πάλι. Δεν ακούγεται. Καλή ιδέα αυτή. Καλό. Τι να κάνουμε λοιπόν. Πολύ καλά. Μόνο εσείς. Και μετά έγινε κιόλα μόλις το είπατε. Ε, κάποιο θαύμα έγινε. 486 υπέρ. Καταπίπτει. Συγγνώμη. Καταπίπτει. 487 υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίθηκε. 489 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Ψηφίζουμε την 489 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Εντάξει. Ένας από το ΕΛΚ παραπάνω. Λοιπόν, πέρας ψηφοφορία τώρα. Εγκρίθηκε. Δεν χρειάζεται 27. 490 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Να ελέγξουμε Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. 490. Ψηφίζουμε την τροπολογία αυτή. Πέρας ψηφοφορίας. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Εγκρίθηκε λοιπόν. 491 τώρα. 491 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 31. Υπέρ της 31. Όχι, τι λέτε εσείς. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Μου διέφυγε μία. Επαναλαμβάνω, συγγνώμη, 493 πρώτα. Ψηφίζουμε την 493 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τώρα έρχεται η 31. Υπέρ της 31, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστώ για αυτό. 30 τώρα, υπέρ. Κατά. Το σκέφτηκα, όλοι εναντίον θα ήταν. Απορρίφθηκε. 31 τώρα λοιπόν, υπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Ήταν σαφές έτσι. Λοιπόν, να μην ζητάμε έλεγχο. Σαφές το αποτέλεσμα. 494 υπέρ κατά, αποχές εγκρίθηκε. 31 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 32 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 495 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 43 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε τη 43. Πέρας ψηφοφορίας. Ένας από το ΕΛΚ παραπάνω. Εντάξει τώρα. Πέρας ψηφοφορίας λοιπόν. Απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε. 43. Υπέρ. «33, ζητώ συγγνώμη» λέει ο πρόεδρος. Φυσικά μόλις ψηφίσαμε τη 43. 33. υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίφθηκε η 33. Έλεγχος. Εντάξει, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. Απορρίφθηκε σαφέστατα. Μάλιστα. Βλέπω καλά. <laughs> Ακόμα και το πρωί. Συμβιβασμός 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε 44 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 45 45 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε καταπίπτει αυτή 47 καταπίπτει τροπολογία 1 του εισηγητή υπέρ υπέρ της 1 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 49 υπέρ καταπίπτει συγγνώμη εντάξει καταπίπτει και η άλλη τροπολογία 2 τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 1 της ΕΚΟΝ Οικονομικής Επιτροπής υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πόσες φορές θα έχουμε την τροπολογία ένα πρόεδρε, είναι πάντα διαφορετική. Αυτή είναι της Επιτροπής Οικονομικών. Εντάξει, συνάδελφε, ωραία. Ε, δεν θα μπορούσαμε να τις διαφοροποιούμε με κάποιο τρόπο θα λέω πάντα ένα, αλλά αυτή τη φορά της Οικονομικής Επιτροπής. Με επιθυμία του συναδέλφου θα υπεξηγώ για ποια τροπολογία ένα πρόκειται εκάστοτε. 54 υπέρ. Κατά. Να επαναλάβουμε. Υπέρ της 54. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. τοπολογία 1 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Ένβη Έλέγχο στην 54, εντάξει, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε την 54. Πέρας ψηφοφορίας. Δύο είπατε, δύο παραπάνω από το ΕΛΚ. Ε, πολλαπλασιάζονται οι του ΕΛΚ. Και χαίρομαι γι' αυτό, για το ότι πολλαπλασιάζονται, αλλά Συγγνώμη, δεν επιτρέπεται να το πω αυτό, ε. Εντάξει. Ωραία. Αμερόληπτος λέει ο πρόεδρος. Πολύ ωραία κύριε Τούρμες. Ναι, πρέπει να τηρούμε τους κανόνες, έχετε δίκιο. Συγγνώμη. Ένας παραπάνω πάλι από το ΕΛΚ. Ένας από το ΕΛΚ παραπάνω. Εντάξει λοιπόν, ρυθμίστηκε. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Τροπολογία 1 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Καταπίπτει, ωραία. Καταπίπτει και η άλλη και η παρακάτω που φτάνουμε 59. Τι λέτε την δύο. Οι δύο λοιπόν της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 58 αυτή καταπίπτει όμως 59 καταπίπτει η 60 και αυτή η 60 όμως είναι συμβατή η 60 υπέρ χωρίς μικρόφωνο η παρέμβαση δεν ακούστηκε Λοιπόν, θα ξαναδοκιμάσουμε. Η 59 λοιπόν, αφού είναι 59 του κ. Τσουκαλά, θα ψηφίσουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 61 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 62 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. Τρία τη Επιτροπή Περιβάλλοντο. ΕΝΒΗ. Έλεγχο θέλετε. Εντάξει, όλο και περισσότερο θα διαρκούν οι ψηφοφορίες. 62, Ηλεκτρονικό έλεγχο άρχεται. Πέρας ψηφοφορία. Ένα από το ΕΛΚ παραπάνω. Τι θα γίνει, θα μπορέσετε να το φτιάξετε αυτό, να το ρυθμίσετε. 62, πέρα ψηφοφορία. Αποτέλεσμα. Ένα λεπτό. Λοιπόν, αυτό σημαίνει απορρίφθηκε. Τρία. επιτροπή Περιβάλλοντος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Κατά τι λέει αν εγκριθεί η άλλη. Οι δύο τώρα. Υπέρ τις δύο. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Τρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 4 καταπίπτει, η 3 καταπίπτει. 66, 66 λοιπόν υπέρ α, κατά αποχές απορρίφθηκε. Περνάμε τώρα 67, 68, 69, 70 ταυτόσημες υπέρ αυτών κατά, αποχές εγκρίθηκαν. Η τρία, υπέρ. Τρία, ΙΜΚΟ όμως. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Η τέσσερα, Επιτροπής Εξωτερικών, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Η τέσσερα, ΙΜΚΟ, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Η 73 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 74, 75 και 5 της ΙΜΚΟ. Όχι, 74 και 75 υπέρ αυτών των δύο. 74-75 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκαν. Να ελέγξουμε, πολύ ωραία, ελέγχουμε. 74 και 75. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Και το αποτέλεσμα γίνονται δεκτές, εγκρίνονται. 5 της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Η 6 ΙΜΚΟ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Η 79 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Η 80 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 81 και 82 υπέρ αυτών. Α, καταπίπτει αυτή. Α, εντάξει, αν εγκριθεί τη ΣΥΜΚΟ η τροπολογία. Καταπίπτουν λοιπόν. Περνάμε στην 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίφθηκε. Η 8 τη ΣΥΜΚΟ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 84, 85, 86, 87. Ταυτόσιμες. Υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκαν. Η 6 ένβη υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Οι 88 και 89 αποσύρθηκαν, συγγνώμη λοιπόν. Η 90 τώρα. 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 7 ένβη υπέρ Καταπίπτει. Ωραία. Καταπίπτει, καταπίπτει. 5, 9, 2. Ε, όλες αυτές καταπίπτουν. Ωραία. Περνάμε στην 106. Δεν καταπίπτει αυτή. 106. Ψηφίζουμε υπέρ. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Η 100 υπέρ Καταπίπτει λέτε. Ωραία, εντάξει. Εγκρίθηκε η 106. Περνάμε στην 101, 102 καταπίπτει, καταπίπτει 107, 107. 107 λοιπόν, υπέρ. Α, κατά, α, αποχές απορρίφθηκε. 108, ως προσθήκη, υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίθηκε Τρία έκον υπέρ α, κατά αποχές εγκρίθηκε τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας ένας από το ΕΛΚ παραπάνω πάλι παρακαλώ ένας από το ΕΛΚ τι γίνεται εντάξει ωραία πέρας ψηφοφορίας Εγκρίθηκε λοιπόν. Και περνάμε στο νομοθετικό ψήφισμα. Τελική απόφαση. Ηλεκτρονικά και πάλι έτσι ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Μια στιγμή. Άρχεται η ψηφοφορία και πάλι. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Και αυτό δεκτό το νομοθετικό ψήφισμα. Ευχαριστώ εγκρίθηκε αυτή η έκθεση. Συγχαρητήρια στον συνάδελφο Βιντάκου Άντρας και ευχαριστώ προσωπικά για τις πολλές συμβιβαστικέ τροπολογίες που διευκόλυναν τώρα τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Επόμενη έκθεση, Πιλάντερ Καστίγιο. Περνάμε στην έκθεση Πιλάντερ Καστίγιο. Ψηφιακή πρώτη ψηφοφορία. Συμβιβασμός 1 υπέρ του, της συμβαστικής τροπολογίας 1. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Ήμκο 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε ΙΜΚΟ 15 ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβασμός 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 106. 106 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 108, 109, 110 σημαίνει υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκαν. Συμβιβασμός 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 127 υπέρ κατά, αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 139 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Τώρα 140, 141, 142, 143, 44, 45, όλες ταυτόσημες υπέρ αυτών. Κατά, αποχές εγκρίθηκαν 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβασμός 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβασμός 10 υπέρ Θέλετε για το 10. Τι. Ε, μια στιγμή, μια στιγμή. Θέλατε να πείτε κάτι για τη 10. Κοιτάξτε, στο συμβαστική 10 θα ήθελα η τροπολογία 166 να ψηφιστεί ξεχωριστά ή δυνατόν. Να ψηφίσουμε ξεχωριστά την τροπολογία 166. Ah, that comes to number 13 later. Okay. Ε, εντάξει. Λοιπόν, θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό υστερότερα σε αυτό το θέμα και θα το διευθετήσουμε. Συμβιβασμό 10. Ψηφίζουμε υπέρ. 10 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίθηκε. 11 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίθηκε. Τώρα. Επιτροπή Πολιτισμού. 19 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίθηκε. Κουλτ 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τι έχουμε τώρα, καταπίπτει, 168 καταπίπτει. Πιλά, Πιλάτα Καστίγιο, τι λέτε. Δεδομένου του κατάλογου ψηφορία, κοιτάξτε, ε, πρέπει να φροντίσουμε, να προσέξουμε λίγο, γιατί πάμε πολύ γρήγορα. Ε, είναι πολύ δύσκολο να τα βλέπουμε όλα αυτά αμέσω. Ε, Σα παρακαλώ, αν θέλετε, ε, λίγα δευτερόλεπτα περισσότερο να μας δίνετε, λίγο πιο ήρεμα. Γιατί διαφορετικά δεν χανόμαστε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποια τροπολογία ψηφίζουμε. Σας παρακαλώ λοιπόν αν έχετε την καλοσύνη. Ναι, αλλά πού υπήρξε το πρόβλημα, σε ποιο σημείο δημιουργήθηκε πρόβλημα, δεν το κατανοώ. Ψηφίσαμε την 19 και είπαμε τη ε, επιτροπή Πολιτισμού που εγκρίθηκε εντάξει η τρία της Επιτροπής Πολιτισμού. Ε, ε, το μόνο που σας ζητώ είναι να πηγαίνουμε λίγο πιο αργά. Όταν κάνουμε αυτά τα άλματα και πηδάμε σελίδε, πρέπει να, να βλέπουμε ποια τροπολογία ψηφίζουμε. Επειδή πολλέ φορέ, όπω σα είπα, κάνουμε αυτό το άλμα και πάμε πολλέ σελίδε παρακάτω, δεν προλαβαίνουμε. Εντάξει, σα ευχαριστώ. Θα επιβραδύνω λίγο. Έλπιζα και νόμιζα ότι θέλατε να τελειώσουμε πιο γρήγορα. Αλλά εντάξει, πρέπει να γίνουν τα πράγματα σωστά. Θα προσπαθήσω λοιπόν τώρα. Charles και πάλι διαδικαστικό. Ε, ε, ε, Πρόεδρε, μας είπατε ότι ήταν η 13 του πολιτισμού. Οπότε εκεί ίσω να δημιουργήθηκε σύγχυση, γιατί ήταν πολιτισμού 3 στον κατάλογο. Ίσως να υπήρξε κάποια παρεξήγηση. Λοιπόν, είχαμε την 19 της Επιτροπής Πολιτισμού και την 3 της Επιτροπής Πολιτισμού και την 168 της κυρίας Ρης που καταπίπτει όμως, καταπίπτει Θλιβόμαστε βέβαια ή οτιδήποτε, αλλά καταπίπτει. Περνάμε στην, συμβαστική 12. Να μην κάνουμε, μην τα μπερδεύουμε πάλι. Λοιπόν, ψηφίζουμε το συμβασμό 12. Υπέρ. Κατά. Ναι, μετά αυτό. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, εγκρίθηκε ο σύμβασμος 12. Περνάμε τώρα στην 173. Τροπολογία 173 υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτή εγκρίθηκε. Και τώρα ο συνάδελφος Σένσο παρακαλώ. Κάντρου κομπρομίσου 13 κα αφορά την συμβαστική 13 θα ήθελα η τροπολογία 166 να ψηφιστεί ξεχωριστά για τους λόγους που εξήγησα χθες το βράδυ ε, τότε να απευθύνουμε ερώτημα προ την εισηγήτρια και στου κοιόδης εισηγητέ. Εντάξει, γίνεται, συμφωνείτε. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Er λοιπόν, συμβιβασμό 13 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίθηκε. Και τώρα η 166 ξεχωριστά όπω ζητήθηκε από τον κύριο Εντσού. Ποιοι είναι υπέρ, Εντσού, 166. Ξεχωριστά θα ψηφιστεί Εντάξει. Μπορούμε να ε, έχουμε προβλήματα τώρα με αυτό, γιατί δεν έχει σημειωθεί στον πίνακα. Λοιπόν, σας αφήνω να το σκεφτείτε λίγο και να διαβάσετε ξανά ίσως την τροπολογία αν θέλετε. Τώρα ψηφίζουμε όμως 166 υπέρ. Κατά αποχές ε, εντάξει με μεγάλη πλειοψηφία 179 ξεχωριστά σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά απορρίφθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε της Επιτροπής Πολιτισμού 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Επιτροπή Πολιτισμού 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Συμβιβασμός 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Ξεχωριστή ψηφοφορία. 202 τροπολογία υπέρ. η 200 καλύπτεται από το συμβιβασμό σύμφωνα με την άποψη τη της, εισηγήτριας. 202 τώρα υπέρ. 202 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 201 υπέρ. Α, καταπίπτει. Ωραία. Καταπίπτει. Επειδή 202 εγκρίθηκε πιο πριν. Περνάμε στο συμβιβασμό 17 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Συ... Όχι, 220 εκ, ξεχωριστά, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 233 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 21. Συμβιβασμός 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 22. Όχι, όχι, ε. Α, ιστερότερα. <laughs> ο συμβιβασμός αυτός. Η 253 τώρα. 253 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 254 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ήμκο 10 τώρα. Η 10 της Ήμκο υπέρ κατά. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 10 της ΣΥΜΚΟ ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Και το αποτέλεσμα γίνεται δεκτή, εγκρίνεται. Η τέσσερα της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Η πέντε της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Η 12 και η 15 της Επιτροπής Πολιτισμού ομού υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκαν οι 6 της Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Οι 275 Βέμπερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 277 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 14 Επιτροπής Πολιτισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Οι 278 και 278 και 283 ομού υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκαν. Έλεγχος, πολύ καλά. 278 και 283 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας και το αποτέλεσμα είναι απορρίφθηκαν. 280 υπέρ. Α, εντάξει, 279. 279 γκρότε υπέρ. Κατά. Αποχές. Παρέμβαση εκτός μικροφώνου. Και πάλι πείτε ξαν Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε. 279. 279 και πάλι υπέρ κατά, αποχές, απορρίφθηκε παρόλα αυτά. 280 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 281 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 282 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Καταπίπτει άλλη 107 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 284 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 285 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 287 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 288 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 23 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε 287 υπέρ κατά αποχές 299 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε της Επιτροπής Πολιτισμού 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 300 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 301 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβασμός 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβασμός 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβασμός 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ξεχωριστή ψηφοφορία, τροπολογία 11 υπέρ, κατά <clears throat> αποχές εγκρίθηκε. 27, συμβιβασμός 27 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 21 καταπίπτει. Καταπίπτει. Ευχαριστώ που μου το είπατε. 21 καταπίπτει. Πολύ καλά. Συμβιβασμός 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 33 υπέρ κατά αποχές και αυτή εγκρίθηκε 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 36, 37, 38, 39 και 40 και 40 ταυτόσημες υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν. Συμβιβασμός 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 44 όχι καταπίπτει αυτή. 45 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε τη 45. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Και το αποτέλεσμα απορρίφθηκε. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. Όχι. Παρακαλώ, 46 και πάλι, υπέρ. Νομίζω ήταν η πλειοψηφία. Κατά, αποχές, μάλιστα, εγκρίθηκε λοιπόν. 49, υπέρ. Κατά, αποχές απορρίφθηκε 50 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 1, 2, 3 καταπίπτουν Α, πρέπει να ψηφίσουμε το κείμενο όπως είχε οτροποποιηθεί τροποποιηθεί όπως είχε δεν το είχα σκεφτεί πιο πριν λοιπόν ηλεκτρονικά τώρα Μόνο τροπολογίες. Όχι ηλεκτρονικά. Λοιπόν, εντάξει, θα ψηφίσουμε έτσι, σηκώνοντα το χέρι. Ποιοι είναι υπέρ του κειμένου ως έχει. Να σηκώσετε το χέρι, παρακαλώ. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτό πρέπει να κάνουμε. Κατά. Αποχέ. εγκρίθηκε το κείμενο. Τώρα περνάμε τώρα. Παρακαλώ, εσείς τι λέτε. Κύριε Πρόεδρε, ε, στην, στη σκέψη 5, τροπολογία 5 δεν την ψηφίσαμε. Θα φτάσουμε σε αυτή. Θα το κάνουμε τώρα. Θα ψηφίσουμε τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, περνάμε, λέει ο πρόεδρο, στι πρόσθετες τροπολογίες. Αυτές είναι για το ψήφισμα. Η 1, η 2 και η 3. 1, 2 και 3 από κοινού ταυτόσημες υπέρ αυτών κατά εγκρίνονται, εγκρίνονται. Τέσσερα. Ακαταπίπτει αυτή. Η πέντε τώρα. Η πέντε υπέρ. Κατά. Η πλειοψηφία, έτσι. Εντάξει, εγκρίθηκε. Ε, συγγνώμη, απορρίφθηκε λέει ο πρόεδρος. Απορρίφθηκε, μάλιστα. Απορρίφθηκε. Έλεγχος ζητάτε. Εντάξει, έλεγχος. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 5. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Και το αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Και το αποτέλεσμα... Εξαιρετικό αποτέλεσμα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια κυρία Πιλάντερ Καστίγιο και ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνατε. Ευχαριστώ θερμά επίσης και για το ότι διευκολύνθηκε η εργασία με τις συμβαστικέ τροπολογίες. Περνάμε στην έκθεση του κυρίου Ρόμπερτ Γκλάντε, Νόρμπερτ Γκλάντε, με συγχωρείτε. Νόρμπερτ Γκλάντε. Θα ήθελα να πει δύο λόγια πιο πριν, πριν ψηφίσουμε ο κύριος Γκλάντε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ σύντομα μόνο. Θα ήθελα ρητά να ευχαριστήσω τους συνεργάτες και συνεργάτριες φυσικά όσον αφορά την Επιτροπή και την Επιτροπή, Επιτροπή, μας, Επιτροπή Προϋπολογισμών και τις ε, εμπλεκόμενες ε, ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές και τους εισηγητές. Είχαμε και συμφωνη, συντονιστεί για την τροπολο, τις τροπολογίες σε σχέση με την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ζητώ συγγνώμη για το ότι έγινε το τελευταίο λεπτό αυτό. Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους, αλλά θέλαμε από τα κονδύλια για τον προϋπολογισμό να αντλήσουμε ό,τι γινόταν παραπάνω. Και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για τον, την τελική χρήση χρηματοδότηση, διότι υποχρηματοδοτήθηκε αυτό το σχέδιο και ελπίζουμε ότι μπορεί να επιτευχθεί αυτή η αύξηση χρηματοδότησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά Νόμπερ Λάντε και για αυτές τις διαπραγματεύσεις που κάνατε. Περνάμε στις ε, τροπολογίες. nv Envy1, υπέρ. Κατά. Να επαναλάβουμε παρακαλώ. Ίσως μπορείτε να με βοηθήσετε λίγο. Συνεχίζουμε έτσι, έχουμε πολλές τροπολογίες. NV1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την NV1. Πέρας ψηφοφορίας. Αρκετοί από όλους. Δεν υπάρχει κανείς παραπάνω. Εντάξει, εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε λοιπόν. 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 26 υπέρ κατά αποχές και αυτή εγκρίθηκε. Περνάμε στην 27. Σωστό. Ωραία. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 29 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 7 και 8 ομού υπέρ αυτών, κατά, αποχές εγκρίθηκαν. Συμβιβασμός 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Τώρα συμβιβασμός 2 και συμβιβασμός 7 ομού υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν οι δύο συμβιβασμοί. Περνάμε στην 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ένβη, η Ενβι 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 11 και της Επιτροπής Προϋπολογισμών 6 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν. Συμβιβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Σε ξεχωριστή ψηφοφορία 42 πρώτο τμήμα υπέρ. Δευ... Συγγνώμη κατά. Να ελέγξουμε. Πρώτο τμήμα της 42. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας ένας σοσιαλιστής παραπάνω στην ψηφοφορία. Διευθετήθηκε τώρα. Ένας παραπάνω είπαμε. Ωραία. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Και το αποτέλεσμα εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 14. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. <clears throat> Της Επιτροπής που είναι 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 45 Κατά πίπλη λέτε. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 17. 17 πρώτα υπέρ. Πρώτα η 17 εντάξει. Η 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Προϋπολογισμό 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Προϋπολογισμόν 1, πρώτη παράγραφος, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 9, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Συμβασμός 10. Όχι, συγγνώμη. Η τροπολογία 2 πρώτα. Τροπολογία 2, 2 του συγητή υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 10. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στην 24. 24 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 5 εγκρίθηκε η τροπολογία και καταπίπτει. Τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Όλα εντάξει. Οκ, λοιπόν. Πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα. Εγκρίθηκε. Κανένα πρόβλημα. Συγχαρητήρια κύριε Γκλάντε λοιπόν. Νομοθετικό ψήφισμα. Και δεν έχουμε νομοθετικό ψήφισμα σήμερα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά οι διαβουλεύσεις για την έκθεση της κυρίας Σαρτόρη και εδώ έχουμε μεγάλο κατάλογο τροπολογιών. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με το συμβασμό 1 υπέρ. Συγγνώμη όμως πρώτα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω το εξή. Μετά από μια ε, συμφωνία με την εισηγήτρια, θέλω να αποσύρω από την ε, τροπολογία 99 το δεύτερο μέρο. Θέλετε να διαβάσω το ε, σημείο αυτό, πάντω είναι σε συμφωνία με την εισηγήτρια. Λοιπόν, όταν θα έρθει η ώρα για να ψηφίσουμε, η 99 αποσύρεται, σημειώνεται. Αποσύρθηκε η 99, να το θυμηθούμε όταν θα έρθει η ώρα λοιπόν. Ωραία, δεύτερο, το δεύτερο τμήμα. 99, 99. Merci, bonjour. <laughs> Also, Kompromiss 1. Λοιπόν, συμβασμό 1. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίθηκε. 65 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίθηκε. 69 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 70 ο καταπίπτη. Μάλιστα, καταπίπτη. 73 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίθηκε. 74 καταπίπτη, 72 καταπίπτη, 10 τώρα υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμό 2 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίθηκε. 77 υπέρ κατά ναι, 77 είπαμε, 77. 77 καταπίπτει, τι λέτε, η 77 καταπίπτει γιατί. Όχι. Ερώτηση. Η 77 καταπίπτει ή όχι. Όχι λοιπόν. Ωραία. Καθόλου. Πολύ σωστό. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε την 77. Ε, καμιά φορά έχουμε και δίκιο. 77 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 78, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 12, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 79 καταπίπτει, η 80, η 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Καταπίπτει άλλη 100 καταπίπτει. 88. 88 υπέρ κατά αποχές υπέρ και πάλι. 88 υπέρ. Υπέρ 88 και πάλι 88 υπέρ Κατά. Εντάξει, εγκρίθηκε. Η 89 καταπίπτει ή 90. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 91 καταπίπτει, 93 καταπίπτει, 94. 94 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Η 17 Διευθετήθηκε η 95 υπέρ. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 97 καταπίπτει 96. 98. 98 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 99. Μόνο το δεύτερο τμήμα της 99. Χωρίς το δεύτερο τμήμα. 99 λοιπόν. Χωρίς το δεύτερο τμήμα. Εντάξει, αυτό θα γίνει. Σωστό. Ωραία. Ψηφίζουμε χωρίς το δεύτερο τμήμα. Έτσι λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, εντάξει, εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 101 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 20 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 102 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 23 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 24 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε 103 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε διαμαρτυρίες τι είπατε 103 ήτανε αποσύρθηκε όχι κύριε όχι απορρίφθηκε το ίδιο δεν είναι ή απορρίφθηκε ή αποσύρθηκε συγγνώμη για το σχόλιο Λοιπόν, 25. Αν είναι τόσο σημαντικό, ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι εντάξει αποσύρθηκε έστω, 20, έστω 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε, 104 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε, 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε, 105 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε, Καταπίπτει, καταπίπτει. Άλλη 107 υπέρ. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 109 υπέρ. 109 είπαμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε.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 κατά αποχές εγκρίθηκε 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 40 ως προσθήκη. 40 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 41 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 42 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Οι 2 τώρα. 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 43 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε 44 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε 45 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε 46 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε 47 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε Τέσσερα. υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε η τέσσερα απορρίφθηκε. Να ελέγξουμε. Ωραία. Έστω. Ελέγχουμε. Ψηφίζουμε την τέσσερα ηλεκτρονικά. Εγώ νομίζω ότι απορρίφθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Εντάξει. Πέρας ψηφοφορίας. Και το αποτέλεσμα ε, υιοθετήθηκε, εγκρίθηκε, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Η 4 εγκρίθηκε λοιπόν, 48 διευθετήθηκε, η 49 ως προσθήκη, έτσι. 49 ως προσθήκη, υπέρ. Κατά. Λοιπόν, θα πρέπει όλοι να συμμετέχουν, να σηκώνετε τα χέρια. Και πάλι, 49, υπέρ. Παρακαλώ. Ε, σαφώς, σαφές το αποτέλεσμα. Εγκρίθηκε. 51 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 52 καταπίπτει. Η, 50, η 53 τώρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 54 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 56 τώρα υπέρ. 56 υπέρ. 56 κατά αποχές εγκρίθηκε 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 5 υπέρ κατά και πάλι λοιπόν 5 υπέρ Σαφές. Εντάξει, διευθετήθηκε. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 60 ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 62 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 63 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Καταπίπτει 64. Τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Ένα σοσιαλιστής παραπάνω όμως. Ένας παραπάνω από τους σοσιαλιστές. Εντάξει τώρα, πέρας ψηφοφορίας. Και το αποτέλεσμα Πολύ καλά, λοιπόν εγκρίνεται. Θερμά συγχαρητήρια κύριε, κύριε, κυρία Σκιώδη συγγήτρια. Μάλιστα. Πολύ καλά, έβγε. Περνάμε, περνάμε στην έκθεση του κυρίου Χατζη Μαρκάκη τώρα. Διαδικαστικό εσείς. Εντάξει συνάδελφε, παρακαλώ. Θα ήθελα να σας ενημερώσω, να σας πω ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα αναβάλει την ψηφορία ε, βάσει του άρθρου 53 του κανονισμού, διότι η Επιτροπή πρόκειται να κάνει νέα πρόταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό η θέση των Πρασίνων θα είναι να καταψηφιστεί αυτή η πρόταση. Okay. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε, λέει ο Πρόεδρος. Κατάλαβα, κατάλαβα. Θα ψηφίσουμε όμως παρόλα αυτά, θα ψηφίσουμε. Ας ψηφίσουμε. 23 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ξεχωριστή ψηφοφορία στην 7 πρώτο τμήμα υπέρ. Εφτά εξαιρείται. Εξαιρείται το κείμενο, μένει εκτός. Νομίζω ότι αυτό, αυτό σας είπα ακριβώς. 7, πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 σαν προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην 27 σε δύο τμήματα σαν προσθήκη. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Επίσης εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 28. Σαν προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. 8 λοιπόν, ε, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33 ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 32 σαν προσθήκη υπέρ. Κατά... κατά αποχές εγκρίθηκε. 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 35 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 36 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 38 το δεύτερο τμήμα δεύτερο τμήμα ως προσθήκη το δεύτερο τμήμα της 38 υπέρ λοιπόν κατά εγκρίθηκε αποχές συγγνώμη εγκρίθηκε ωραία 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 40 δεύτερο τμήμα ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές και αυτό εγκρίθηκε. Περνάμε στις 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε ή 42 υπέρ κατά κατά αποχές εγκρίθηκε. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε περνάμε πίπτη άλλη 46 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 51 υπέρ κατά θα ελέγξουμε ψηφίζουμε την 51 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά 51 εντάξει ελέγχουμε άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας και το αποτέλεσμα απορρίφθηκε 17 υπέρ κατά, αποχές εγκρίθηκε 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβασμός 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 3 χωρίς τη διατύπωση που ακολουθεί εδώ. Λοιπόν, όσοι είναι με αυτήν την τροποποιημένη διατύπωση υπέρ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τέσσερα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 21. Ως προσθήκη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 22. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά ψηφίζουμε άρχεται πέρας ψηφοφορίας μάλιστα εξαιρετικά εγκρίθηκε συγχαρητήρια επόμενη ψηφοφορία κυρίου Χατζημαρκάκη και πάλι Χατζημαρκάκης λοιπόν Έχουμε την 6 της έκθεση Χατζημαρκάκη. Ξεκινάμε με την τροπολογία 6. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Η 7 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Η 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Η 8 Μπορούμε να τις ψηφίσουμε όλες αυτές εδώ στη σειρά, ομού. Μπορούμε ομού να ψηφίσουμε από την 8 στην 1. Εντάξει, γίνεται. Από την 8 στην 1 λέω. Εντάξει, ομού. Όλοι σύμφωνα. Είναι κάποιος εναντίον. Όχι, ωραία. Αποχές κανείς. Λοιπόν, εγκρίνονται όλες αυτές. Τέλεια. Και περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Καλή ιδέα ήταν. Άρχεται η, η ψηφοφορία, τέλος ψηφοφορίας και το αποτέλεσμα Λοιπόν, εγκρίθηκε. Πολύ καλά. Πάει και αυτό. Μεγάλη πλειοψηφία. Και περνάμε τώρα στην ψηφοφορία. Φραντσέσκο Ντε Άντζελης για αυτή την έκθεση. Πάλι πολλές τροπολογίες έχουμε εδώ. Ξεκινάμε με τη 14. Συγγνώμη, κυρία Τούρμες. Ο Κλωτ Τούρμες, συγγνώμη. Δεν λειτουργήσε το μηχάνημά μου, δεν λειτουργήσε. Να βάλετε και εμένα και δική ψήφο κατά. <laughs> Ωραία, λοιπόν, σας ευχαριστώ. Έκτη ψήφος εναντίον να κατατεθεί στα πρακτικά. Έγινε λοιπόν η δουλειά πιο πριν. Πολύ καλά. Φραντσέσκο Ντε Άντζελης, η 14 λοιπόν τροπολογία. Λειτουργεί τώρα Κλοντ. Κλοντ Τούρμες, ποιοι είναι υπέρ της 14. Κατά αποχές, εγκρίνεται. Η 1, 12, 13 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 17 υπέρ κατά τι γίνεται εδώ να ελέγξουμε λοιπόν ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται ψηφίζουμε την 17 ηλεκτρονικά άρχεται Πέρας ψηφοφορίας. Ε, βλέπετε ισοψηφία. Αυτό είναι. Πολύ αργά τώρα όμως. Πολύ αργά λυπούμε. Ψηφίσαμε ήδη. Τελειώσαμε. Τι λες εσύ, τι έχεις. Δεν λειτουργούσε με την κάρτα σου. Κλοντ, το ίδιο πρόβλημα και εσύ. Λοιπόν, τι, πώς ήθελες να ψηφίσεις εσύ ή να υπερψηφίσεις και εσείς να καταψηφίσει; Ε, δεν αλλάζει τίποτα. Τέλεια. Ωραία. Πολύ καλά. Πρωτότυπο αυτό. Να καταχωρηθεί στις ιστορικές δέλτους των ψηφοφοριών στην Ευρωβουλή. Ε, παρόλα αυτά απορρίφθηκε. Λοιπόν, τι κρίμα. Απορρίφθηκε. Περνάμε στο συμβιβασμό 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίθηκε. Θεέ, να προσέξουμε τώρα εδώ. Η τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 24 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 25 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 52 52 υπέρ 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 54 ως προσθήκη υπέρ κατά Να ελέγξουμε λοιπόν. Ψηφίζουμε την 54 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Έτσι. Εγκρίθηκε. Κλοντ, τι έγινε με σένα. Ναι, πώς ήθελες να ψηφίσεις, τι ήτανε. Πώς υπεψηφίζεις ή καταψηφίζεις. Α, λειτουργεί τώρα η συσκευή σου. Πολύ καλά. Λοιπόν, τέλεια. Λειτουργεί. Εγκρίθηκε λοιπόν. Ας μην δώσουμε συνέχεια εδώ. 56, 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στην 55 που την ξεχάσαμε. 55 λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές και αυτή εγκρίθηκε. Τώρα περνάμε στην 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 57 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε και περνάμε στην 11 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται όλα εντάξει όλα εντάξει Πέρας ψηφοφορίας. Και το αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια. Και πάλι τώρα Χατζημαρκάκης εδώ στην ψηφοφορία. Χατζημαρκάκης άλλη μια φορά. Τι γίνεται δεν λειτουργούν συσκευές, τέλος πάντων. Ξεκινάμε με το συμβιβασμό 1. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε σε ξεχωριστή ψηφοφορία για το 3. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 3. Δεύτερο. Υπέρ. Κατά αποχές και αυτό εγκρίθηκε. τέσσερα τώρα, τροπολογία τέσσερα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός επτά υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Το συμβασμός έξι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός, συμβιβασμός 5, όχι, Α, συγγνώμη. Μάλιστα. τρία. Συμβασμός τρία Στο τέλος της γραμμής αυτή. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβασμός πέντε Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Συμβασμός δύο Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16. Ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία ψηφίζουμε την 17 17 λοιπόν 17 άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας και το αποτέλεσμα εγκρίθηκε και η 19 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε μάλιστα απορρίφθηκε τι έχουμε εδώ 18 πρώτο τμήμα 18 18 πρώτο τμήμα έτσι ολόκληρη 18 πολύ ωραία ποιοι είναι υπέρ της 18 The vote is 18, number 18. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε και 27 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 28 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε μάλιστα. Και περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Θε. Πάλι. Ωραία. Ομόφωνα. Εγκρίθηκε ομόφωνα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Επόμενη ψηφοφορία. Έκθεση Paul Rubich εδώ η κυρία Τίκα, ο συνάδελφος, ζήτησε πιο πριν δύο-τρία λεπτά να πει κάτι. Η κυρία Τίτσαου έχει τον λόγο για την έκθεση Να πει κάτι παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα έχω προφορική τροπολογία, όπως είπα και χτες, για την τροπολογία μου υπαριθμών 6. Θα διαβάσω την ε, τροπολογία όταν φτάσουμε εκεί και θα παρακαλούσα τους συναδέλφους να μην υποστηρίξουν την αρχική παράγραφο 2 διότι η αδειοδότηση που βασίζεται στις γλώσσες θα είναι κάτι πολύ παρακινδυνευμένο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς εξολόγηση συνεπιών. Και αντί να έχουμε μία άδεια για ένα έργο, θα έπρεπε να έχουμε 23 τουλάχιστον άδειε βάσει γλωσσών. Διότι έχουμε 23 επίσημες γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω οι συνάδελφοι να μην υποστηρίξουν την παράγραφο 2. Θα διαβάσω τη δική μου τροπολογία 6, προφορική τροπολογία όταν φτάσουμε εκεί. Εντάξει, ο Παύλ Ρούμπιχ θα λάβει τον λόγο, παρότι δεν ανοίγουμε συζήτηση τώρα. Εντάξει, δεν το επιτρέπει η διαδικασία. Κύριε Ρούμπιχ, ευχαριστώ Πρόεδρε για αυτό το θέμα που ζητήσαμε την κυρία Σιώδη Συγήτρια Τιτσάου για την τροπολογία της που θα ήταν αποδεκτή αν θα ήταν ξεχωριστή νέα παράγραφος. Είμαστε όμως κατά την δική μας παράγραφο 2 να την τροποποιήσει. Η παράγραφος 2 σε σχέση με τους Ευρωπαίους πολίτες λέει, ότι έχουν το δικαίωμα στα 27 κράτη-μέλη να ακούνε αυτό το περιεχόμενο αυτών των παρεμβάσεων στη δική τους γλώσσα, να το έχουν στη δική τους γλώσσα. Είναι σημαντικό να είναι αυτό το δικαίωμα έτσι. Ευχαριστώ. Περνάμε στην ψήφιση τροπολογία 1 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε τροπολογία 6 η κυρία Τιτσάου είχε προφορική τροποποίηση το κείμενο της προφορικής τροπολογίας τροπολογία παριθμών 6 με την προφορική τροπολογία θα είναι το εξή κείμενο και θα αντικαταστήσει την παράγραφο υπαριθμών 2 θεωρεί σαν ένα βήμα προς εσωτερική αγορά για το IPR μέσα όπως υποτίτλους που προσφέρει ψηφιακή τηλεόραση που δίνει δυνατότητα τη διανομή ενό έργου σε αρκετέ γλώσσε, καθώ και την πρόσβαση του καταναλωτού σε αυτό το έργο στην πρωτότυπη γλώσσα. Και ελπίζω όλοι οι συνάδελφοι να υποστηρίξουν αυτή την τροπολογία. Ευχαριστώ θερμά. Λέει ο Πρόεδρο, υπάρχουν ενστάσει, αντιρρήσει για αυτή την προφορική τροποποίηση. Ο κύριο Πίτερ Χόφερ, παρακαλώ. Πρόεδρε, η συνάδελφο μόλι είπε ότι αυτή η προφορική τροποποίηση θα πρέπει το, την παράγραφο 2 να την αντικαταστήσει. Όμως εμείς έχουμε εγκρίνει το 2. Πώς έχει. Την τροπολογία 2 εγκρίναμε λέει ο Πρόεδρος. Εδώ πρόκειται όμως για την παράγραφο 2. Εντάξει και εγώ είχα ε, κάποια αμφιβολία αλλά μόλις το είδα και έτσι είναι. Λοιπόν συμφωνείτε. Λοιπόν ε, δεκτή η τροποποίηση, ψηφίζουμε την τροποποίηση συναδέφου ΤΙΚΑΟ και έτσι πάει η τροπολογία 6. Προφορική τροποποίηση ΤΙΚΑΟ υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Επτά τώρα υπέρ να ελέγξουμε ωραία προφορική τροποποίηση ελέγχουμε άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά τέλος ψηφοφορίας και το αποτέλεσμα απορρίφθηκε μάλιστα πολύ καλά Επτά τώρα τροπολογία επτά. υπέρ Παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο. Δεν ακούστηκε. Τι είπατε. Okay. Ah, Πολύ καλά. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, την προφορική τροποποίηση την είχα κατανοήσει ότι αντικαθιστούσε την τροπολογία 6, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Η 6 Θέλει η συνάδελφο να ψηφιστεί και αυτή ξεχωριστά. Ψηφίζουμε φυσικά την τροπολογία 6 της κυρίας Τίκαου ξεχωριστά. Η κυρία Τίκαου ήθελε σε σχέση με την 6 να ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε την 6 της κυρίας Τίκαου. Υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ αυτής της τροπολογίας. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε την αρχική τροπολογία. Την αρχική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Τώρα αυτή εγκρίθηκε. Και τώρα περνάμε στην 7. 7 λοιπόν υπέρ. Ωραία. Πολύ καλά, εντάξει. Θα ελέγξουμε και για το 2 το τμήμα 2 στην αρχική διατύπωση. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ελέγχουμε. Πέρας ψηφοφορίας και το αποτέλεσμα εγκρίθηκε. Και περνάμε στην 7, 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 10 σε τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα της 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα της 10 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε αυτό το δεύτερο. Περνάμε στο συμβιβασμό 1. Έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της 10. Έλεγχος. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία και πάλι. Πέρας ψηφοφορίας. Και το αποτέλεσμα απορρίφθηκε το δεύτερο τμήμα της 10. Περνάμε στο συμβιβασμό 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Η 16 τώρα. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα της 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα της 16. Υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 17 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 19 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε προφορική τροποποίηση τώρα στην παράγραφο, παράγραφο 7α σωστό σωστό το κείμενο το έχετε γραπτά μπροστά σας ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 25 υπέρ 25 όχι καταπίπτει 27 λοιπόν 27 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 26 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 28 υπέρ να ελέγξουμε λέτε πολύ καλά 26 λοιπόν ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Και το αποτέλεσμα εγκρίθηκε 26. Σας ευχαριστώ για αυτό. Δεν το είχα προσέξει. Ευχαριστώ πολύ. Και περνάμε τώρα στην 28. 28 υπέρ. Υπέρ της 28 κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 30 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 31. Όχι, να ελέγξουμε την 30. Πολύ καλά, καλύτερα. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 30. Άρχεται. 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Εντάξει όλα. Και τέλος ψηφοφορίας απορρίφθηκε. Η 31 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Εντάξει. Απορρίφθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίζουμε την 31 ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας Πέρας ψηφοφορίας και το αποτέλεσμα απορρίφθηκε. Τελική ψηφοφορία τώρα ηλεκτρονικά άρχεται. Δεν είχε λέει αναφερθεί το αποτέλεσμα. Δεν αναφέρθηκε στην οθόνη το αποτέλεσμα, λέει. 22-24 το αποτέλεσμα, μάλιστα. 22-24. Τελική ψηφοφορία τώρα, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας και εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο συνάδελφος Βίντα Κουάντρα ζήτησε τον λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα ζήτημα από της διαδικασίας πριν την τελευταία ψηφοφορία. Θα ήθελα να δούμε με τη γραμματεία το εξής κατά πόσο ο αριθμός ε, των τελικών ψήφων στην τελική ψηφοφορία της έκθεσης ε, ε, για την ασφάλεια εφοδιασμού σε φυσικό αέριο ήταν αυτός που έπρεπε ή υπήρχε άλλη μία ψήφος. Θα κάνουμε την επαλήθευση για με ονομαστική ψηφοφορία, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να δούμε κατά πόσον έχουμε υπέρβαση. Το λέω αυτό, Πρόεδρε, γιατί ε, στην περίπτωση των μία γεγραμμένων ψήφισαν τρει και από ό,τι κατάλαβα έχουν δικαίωμα μόνο σε δύο ψήφους στην Επιτροπή. Λοιπόν, ψήφισαν δύο μόνιμα μέλη και ένας ελπιματικός. Και πιστεύω ότι η ομάδα των μία γεγραμμένων πρέπει να ανακοινώσει στη γραμματεία ποια ψήφα αποσύρει, έτσι ώστε η τελική ψηφοφορία να αντικατοπτρίζει πιστά τη θέση τη επιτροπή μα. Πολύ καλά. Εγώ όμω λέω, συνάδελφοι Βιντάρ προσέξτε. Βιντάρ ακούστε. Με, σε κάθε ψηφοφορία ρωτάω πάντα αν είναι ορθός αριθμός ε, των μελών παρόντες ε, και συμμετέχουν στην ψηφοφορία. Υποθέτω ότι αυτό έγινε έτσι. Αν ένας είναι παραπάνω, τότε αυτό θα ελεγχθεί και αν πράγματι συμβαίνει αυτό, τότε θα πρέπει οι ανεξάρτητοι να μας πούν ποιος από αυτούς αποσύρεται, ποιος πιανού η ψήφος θα αφαιρεθεί. Του. Νομίζω ότι μόνο δύο ε, από εμάς είμαστε εδώ, είμαστε πλήρη μέλη εδώ. Δεν ξέρω να υπάρχει άλλος στην αίθουσα. Δεν υπάρχει άλλος μέλος της ομάδας μου εδώ. Okay. Τώρα δεν μπορούμε αυτό να το αποσαφηνίσουμε. Δεν παρενέβη η γραμματεία όταν γινόταν η ψηφοφορία. Δεν μου είπε κανείς ότι ήταν ένας παραπάνω. Αν είναι ένας παραπάνω πρέπει αυτός να αποσυρθεί. Η ψήφος να αφαιρεθεί, να μην συμμετέχει uh, niet ingeschrevenen. Per... Όσον αφορά το θέμα αυτό, θέλω να πω ότι ψήφισα την πρόταση αυτή. Στο τρίτο σημείο δεν... Αποσύρω την ψήφα μου, δεν κατάλαβα ότι ήμασταν τρεις παρόντες, έκανα λάθος. Ευχαριστώ για αυτή την επισήμαση και την αποσαφήνιση διευκολύνει αυτό τα πράγματα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ και ε, όσον αφορά τα πρακτικά, σας παρακαλώ να αναγραφεί ότι, ότι η ψήφος υπέρ της έκθεσης ήταν ομόφωνη. Ευχαριστώ. Εντάξει, θα ελέγξουμε το αποτέλεσμα. Θα αφαιρεθεί η ψήφο του παραπάνω και αντίστοιχα το αποτέλεσμα θα είναι πλέον το επίσημο αποτέλεσμα πια. Εντάξει, σαφέ. Επόμενη ψήφος. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε. Έχετε εσείς προφορική τροποποίηση, κυρία, παρακαλώ. Πρόεδρε, να σας ειδοποιήσω. Θα ήθελα προφορική τροπολογία όσον αφορά την ε, τροπολογία 24. Θα σας δώσω το λόγο όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, λέει πρόεδρος. Πρόεδρε, ah, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, στην επόμενη σύνοδο που θα γίνει η ψηφοφορία μπορούμε να επαληθέσουμε αυτά που κάνατε στην αρχή ε, κατά ομάδα τι έγινε στην Επιτροπή. Διότι περάσατε τον ίμιση χρόνο ε, λέγοντας υπάρχει ένα μέλος του ΕΛΚ παραπάνω, υπάρχει ένα σοσιαλιστής παραπάνω. Να κάνουμε κατά ομάδα επαλήθευση και να γνωρίζουμε αν υπάρχουν αρκετές ψήφοι ή όχι αρκετές ψήφοι, να γίνεται επαλήθευση και έτσι να είμαστε ήσυχοι. Λοιπόν, άλλη μια φορά, σε κάθε ψηφοφορία, σε κάθε ψηφοφορία που στο τέλος γίνεται και ηλεκτρονικά η γραμματεία, ο επικεφαλής γραμματείας ο ίδιος θα κοιτάζει αν σε αυτό τον πίνακα ψηφοφορίας όλα είναι καλά, βαίνουν καλώς και θα μου λέει αν κάποιος είναι παραπάνω και τότε πρέπει να υπάρχει διόρθωση, επανόρθωση. Τότε μόνο. Πιο πριν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί οι συνάδελφοι μπαίνουν, βγαίνουν στην αίθουσα, αλλάζουν τα πράγματα. Δεν είναι πάντα ότι όλοι από τις 9.30 ε, από τις 9 στις 12.30 είναι εδώ παρόντες όλοι. Αλλάζει η σύνθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας της συνεδρίασης. Και εμείς είχαμε πει ότι αυτό ήταν σωστό. Τώρα, ευτυχώς ε, ανακαλύφθηκε το λάθος, αναφέρθηκε, διορθώθηκε και νομίζω αυτή είναι η σωστή διαδικασία. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει. Έγινε η διόρθωση λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για την επισήμανση. Περνάμε τώρα στην, στην έκθεση του κυρίου Τσίτσεστερ και ψηφίζουμε. Μετά υπάρχει και προφορική τροποποίηση της κυρίας Χολ, προφορική πρόταση που θα την εξετάσουμε. Τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 4α υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβαθμός 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τώρα πρέπει να τα δούμε. Η τροπολογία 11, Hall, και η προφορική της τροποποίηση εδώ. Όχι, όχι ακόμα. Εντάξει, 11, υπέρ, 11. Κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Η 13, υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε. Η 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 19 υπέρ κατά να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 19 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Προσέξτε εσείς. Να προσέχετε παρακαλώ. Μην έχουμε κανένα παραπάνω. Όλα εντάξει. Όλα εντάξει. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε 22 σε τμήματα πρώτο τμήμα της 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο της 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 24 Τώρα έχουμε την προφορική τροποποίηση της κυρίας Χολ. Παρακαλώ κυρία Χολ. Ευχαριστώ. Η προφορική τροπολογία είναι απλώς η διαγραφή εξαιρετικής, exceptional Οπότε λέει υπογραμμίζει την περιβαλλοντικά ωφέλη το να έχουμε καύσιμα από βιολογικά απόβλητα αντί να λέμε αυτό ότι υπογραμμίζει τις εξαιρετικ... τα εξαιρετικά περιβαλλοντικά ωφέλη, το εξαιρετικά ε, διαγράφεται. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς να πω ότι είναι στο πρώτο τμήμα. Έχουμε ακόμα ξεχωριστή ψηφοφορία για το δεύτερο κομμάτι τη τροπολογία και ω προφορικά τροποποίηθη θα υπερψηφίσω το πρώτο τμήμα. Οπότε θα αλλάξω, θα δεχτώ την προφορική τροπολογία, αλλάζω αυτή τη θέση μου που είχα στον κατάλογο ψηφοφορία. Λοιπόν, με άλλα λόγια, ψηφίζουμε σε δύο τμήματα. Η προφορική τροποποίηση αφορά το πρώτο τμήμα στο οποίο αναφέρθηκε. Ψηφίζουμε πρώτο τμήμα με την προφορική τροποποίηση κυρία Χόλ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 26. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 29 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 30 σε τμήματα ψηφοφορία. Εντάξει, οι 30 σε... Μόνο το πρώτο τμήμα ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ του πρώτου τμήματος στις 30. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Και έτσι περνάμε στην 31 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Και τώρα τελική ψηφοφορία. Καταλήγουμε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Όλες οι ομάδες με σωστή σύνθεση πέρας ψηφοφορίας και το αποτέλεσμα είναι υπεψηφίστηκε 48 υπέρ, ομόφωνα υιοθετείται. Συγχαρητήρια Τζάις Chichester. Έχετε τις καλύτερες ευχές όλων. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και αυτά ήταν σήμερα της πρωινής μας συνεδρίασης ε, το περιεχόμενο. Είχαμε πολλές ψηφοφορίες. Είχαμε εδώ αν θέλετε και την αθλητική αυτή συνεισφορά αθληθήκαμε. Το απόγευμα θα ξανασυναντηθούμε πάλι. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα το απόγευμα έχουμε έκτακτους κατεξαίρεση φιλοξενουμένους. Θα ήμουν πράγματι ευγνώμων αν γινόταν. Ένα λεπτό, ακούστε, προσέξτε. Ένα λεπτό ακόμα. Κάποιοι από εσάς να έρθετε, οι περισσότεροι από εσά να έρθετε στην απογευματινή συνεδρίαση, γιατί θα έχουμε εξαιρετικούς φιλοξενουμένους. Να μπορέσετε να έρθετε λοιπόν. Ευχαριστώ.